Έχει το λόγο η Φεντερίκα Μογκερίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντάς σας για την εκλογή σας. Είμαι βεβαία ότι θα συνεργαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης. Και ένα στοιχείο το οποίο, με το οποίο συμφωνώ απόλυτα αυτό που είπε η φίλη μας, ε, η φίλη μου, η κυρία Φωτήγα, και η κυρία Κοράτσα Μπίλ στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών την Δευτέρα θα έχουμε το θέμα της, ε, της Ουκρανίας ε, και θα θέσουμε το ζήτημα αυτό. Και τώρα να έρθουμε στο θέμα που μας απασχολεί σήμερα και που είναι στην ημερήσια διάταξή μας σήμερα. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η Ευρώπη και η ΕΠΑ ΕΕ συνδέονται από μια παλιά και βαθιά φιλία προσωπικά πάντα. Θεωρώ ότι είπα με μεγάλο σεβασμό και μεγάλη σεβασμό ως μια χώρα όπου μπορεί κανείς να πετύχει ότι θέλει ανεξάρτητος ε, προέλευσης. Μια χώρα ελπίδας, μια χώρα που πραγματοποιούνται τα όνειρα, μια χώρα η οποία ήταν πάντα μεγάλη ακριβώς επειδή πάντα ήταν ανοιχτή και πάντα ήταν πρωταθλήτρια στις ελευθερίες. Ως καλή φίλη λοιπόν τον είπα, πιστεύω ότι η Ευρώπη έχει ένα καθήκον. Έχει καθήκον να είναι σαφής και να επιδείξει σεβασμό. Οπότε τίθεται θέμα διαφωνίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις θεμελιώδεις ε, αρχές. Και σίγουρα διαφωνούμε με την εκτελεστική εντολή του Πρόεδρου των ΗΠΑ που εκδόθηκε στις 27 Ιανουαρίου. Όπως και πολλοί διαφωνούν φαίνεται στις ΕΠΑ και προβλέπετε λοιπόν μια απαγόρευση εισόδου στη χώρα για 90 ημέρες από 7 χώρες. Και προβλέπεται επίσης προσωρινή αναστολή για 120 ημέρες του προγράμματος ε, των ΕΠΑ για την εισαγωγή για την είσοδο προσφύγων. Μέχρι ότου δηλαδή ο Υπουργός Εξωτερικών και Ασφάλειας αναστήλουν αυτή την ε, περίοδο. Και έχουν τεθεί ερωτήματα για το ποιοι πολίτες θα επηρεαστούν από αυτή την απαγόρευση εισόδου. Το Υπουργείο Εξωτερικών τον είπα, διευκρίνησε χθε ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα επηρεαστούν από την απαγόρευση. Ακόμα και να έχουν υπηκότητα σε μία από τις επτά χώρες αυτές που περιλαμβάνονται. Καλωσορίζουμε αυτή την ευκρίνηση, αλλά θα είμαι εντελώς κατηγορηματική ότι αυτό δεν αλλάζει τη συνολική μας εκτίμηση για την εκτελεστική αυτή εντολή. Και διευκρίνησα τις τελευταίες ημέρες ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το θέμα. Κανείς, και επαναλαμβάνω κανείς, δεν μπορεί να αποστερηθεί από, το δικαίωμα του, από τα δικαιώματά του λόγω χώρου λόγω της χώρας στην οποία γεννήθηκε ή από την οποία προ έρχεται ή λόγω εθνοτική ε, προέλευση. Αυτό ισχύει και κατοχυρώνεται στα συνταγματα και τη Ευρώπης και των Αμερική. Αυτό είναι το ποιοι είμαστε, η ταυτότητά μας. Δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε αυτό. Η ευρωπαϊκή μας ιστορία μας ε, διδάσκει ότι γιορτάζουμε όταν ε, χτίζεται μια γέφυρα και πέφτει ένα τείχο. και έχουμε μάθει από την ιστορία μα ότι κάθε ανθρώπινο όν καταρχά και πρωτίστω είναι ένα άτομο με θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα τα οποία δεν μπορούν να υπονομευθούν. Θα ήθελα από προσωπικής άποψης να σας σχολιάσω ότι είναι πραγματικά λυπηρό. Είναι λυπηρό το ότι ακούσαμε ότι αυτή η εκτελεστική εντολή ε, εκδόθηκε 27 Ιανουαρίου, ημέρα μνήμης του ολοκαυτώματος. για τα θύματα των Ναζί και μια ημέρα μνήμης που καταδικάζουμε οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση και υποστηρίζουμε αυτό. Πολλά από τα θέματα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους ε, φεύγουν και διώκονται από τρομοκρατικά καθεστώτα από αυτό της ΔΑΕΣ. Είναι θύματα και πέρα από το γεγονός ότι είναι ε, πρόσφυγες, είναι άνδρες, γυναίκες, παιδιά με ιστορίες, όνειρα, φόβους και βαθύτατες πληγές. Και έχουν πάνω απ' όλα την επιθυμία να οικοδομήσουν ένα μέλλον και για το καλό των δικών τους χωρών και της ασφάλειάς τους, γιατί η κοινωνική ανοικοδόμηση των χωρών τους από αυτούς εξαρτάται. Ας ε, είμαστε λοιπόν σαφείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα απορρίψει τον οποιονδήποτε που ε, δικαιούται διεθνούς προστασίας. Ε, αυτή ήταν και θα είναι η θέση μας. Δεν θα ήταν ούτε δίκαιο, ούτε ηθικό, ούτε και νόμιμο και δεν θα ήταν και προς το συμφέρον μας αν θέλετε γιατί τέτοιου είδου μέτρα θα α, όξιναν την δυσπιστία, τις τριβές μεταξύ των ανθρώπων, των λαών, των εθνών. Και όταν λέω μεταξύ των ανθρώπων, εννοώ και των ανθρώπων μέσα στις ίδιες μας τις κοινωνίες. Και αν με ανησυχούν οι τάσεις που διακρίνω στην Αμερικανική κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν και κάλεσα τον πρόεδρο τον είπα να προσέξει τι συμβαίνει στην ίδια του τη χώρα πρωτίστως. Μόνο με το σεβασμό και τη συνεργασία μπορούμε να είμαστε πιο ασφαλείς. Μόνο με το σεβασμό και τη συνεργασία μπορούμε να διαχειριστούμε τις πολλαπλές κρίσεις που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος. Συνεργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε με τις χώρες που έχουν κρίση και με τις όμορες χώρες τους. Μία απαγόρευση ταξιδιού Μπορεί, μπορεί ενδεχομένως να δώσει μια προσωρινή ψευδέστηση ότι διαχειριζόμαστε κάποιο θέμα, αλλά ουσιαστικά προκαλεί πιο πολύ αγανάκτηση και θυμό παρά ποτέ. Χρειαζόμαστε συνεργασία και όχι να κλείσουμε με φράγματα. Χρειαζόμαστε να βρούμε κοινό τόπο, όχι που απαγορεύουμε το οτιδήποτε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να είναι εταίρος και ισχυρό σημείο αναφοράς για όλες τις χώρες στην περιφέρεια, στην περιοχή, ανεξάρτητα από την θρησκεία των πολιτών του Μπορούν να υπολογίζουν πάνω μας και θα συνεχίσουμε να είμαστε εταίρος και ισχυρό, στενερό σημείο αναφορά για όλου εκείνου στον κόσμο που πιστεύουν στην διεθνή συνεργασία, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί και το μεγαλύτερο δωρετή του κόσμου στην λαό της Συρίας και στις γειτονικές χώρες. Πάνω από 9 δις έχουμε δώσει από την αρχή της συγκρούσεως στη Συρία και έως τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ έχουν συνεργαστεί στενά και στο πλαίσιο του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Γιατί ένα παγκόσμιο ζήτημα χρήζει παγκόσμια ε, αντιμετώπιση και έχουν αναλυθεί δεσμεύσει για να προστατευτούν τα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων και όλων των προσφύγων η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη σε ανα στιγμή να ε, συζητήσει με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ για να συνεχιστεί αυτή η δέσμευση που έχει ξεκινήσει για να συνεχιστούν τα επιτεύγματα που έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια και σήμερα αυτά είναι τα βασικά θεμελιώδη στοιχεία τη ε, πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, από την αλλαγή του κλίματο, η συμφωνία στο Ιράν, από την ειρήνη στο Μεσανατολικό, την υποστήριξή μα ε, στο σύστημα του ΟΗΕ και ένα ελεύθερο εμπορικό σύστημα. Και βάσει αυτών και βάσει αυτής της σαφέστατης ε, ατζέντα θα ε, συνεργαστούμε με την κυβέρνηση των ΗΠΑ με αμοιβαίο σεβασμό. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή οδός, αυτές είναι οι αρχές μας, οι αξίες μας, αυτό είναι και το συμφέρον μας. Και πιστεύω ότι φέρουμε ευθύνη, φέρουμε ευθύνη και προς τους πολίτες μας και προς τους εταίρους μας στην περιοχή και σε όλο τον κόσμο. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς προς τις αρχές μας να επιδείξουμε ηγεσία και ισχύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Αντιπρόεδρο. Περνάμε τώρα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο κύριος Βέμπερ έχει το λόγο. Αξιότιμη πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, το σημαντικό θέμα, οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί είναι όλοι όμω και καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο. Στηρίζουμε την άποψη που μα παρουσίασε σήμερα η κυρία Μογκερίνη, εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμω νομίζω ότι πρέπει να πούμε κάποια ε, περισσότερα ε, πάνω σε αυτό. Εξελέγει δημοκρατικά, σεβόμαστε αυτή την ε, απόψη του Αμερικανικού λαού. Θα πρέπει να συνεργαστούμε μαζί του, θα πρέπει να χτίσουμε γέφυρε. Σίγουρα υπάρχει σεβασμός. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια διαφοροποίηση ο Ντόναλτ Τραμπ λέει ότι θέλει να καταπολεμήσει την λαθρομετανάστευση. Λέει ότι καταπολεμεί την Ισλαμιστική τρομοκρατία. Και στις δύο περιπτώσεις εμάς το ΕΛΚ μας έχει στο πλευρό του. Επίσης υπήρξε στην τηλεφωνική συνομιλία με την Τερέζα Μέη και με την Άγγελα Μέρκελ και λέει ότι είναι υπέρ του ΝΑΤΟ, κύριο Τραμπ. Και αυτά είναι θετικά. Ε, βέβαια, αυτό το οποίο ε, γέρνει, ε, η πλάστικα γέρνει προς ένα άλλο σημείο, γέρνει προς ε, αυτά που έγινε στις τελευταίες τελευταίες Η Αμερική, κυρίες και κύριοι, είναι η χώρα της ελευθερίας. Η ΕΠΑ είναι η χώρα της μετανάστευσης ε, και τώρα υπάρχουν κάποιες ε, υποψίες ε, γενικές και όλα αυτά δεν οδηγούν σε βελτίωση της κατάστασης, οδηγεί σε ένα νέο μίσος. και ο Καναδός που έκανε ο δράση επίδεση στον Καναδά στράφει εναντίον κατά του Τραμπ ξεκάθαρα. Βλέπουμε λοιπόν τώρα έναν Αμερικανό πρόεδρο που θέλει να κόψει και κάποιες συμφωνίες ό,τι αφορά το χάρη με τον Ειρηνικό, το TTIP. Εμεί ε, δεν τα θέλουμε αυτά φυσικά και θέλουμε να υπάρχει εμπορική εταιρική σχέση θα ψηφίσουμε το Φεβρουάριο και θα δώσουμε ένα σαφές ε, μήνυμα. Θα στηρίξουμε τις προσπάθειες ε, της κύρια Μάστρο με Μεξικό, Καναδά, Ιαπωνία ε, και άλλες χώρες για να ενισχύσουμε τις εμπορικέ σχέσεις, γιατί θέλουμε εμπορικέ συμφωνίες. Και για να δώσω και ένα παράδειγμα ακόμη, η ΠΑ είναι και η χώρα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους και ο κύριος Τραμπ τώρα λέει ότι και τα βασανιστήρια είναι ε, αποτελεσματικά. Δεν μπορεί να αναφέρεται αυτή η λέξη βασανιστήρια από το κράτος, γιατί το κράτος γίνεται αμέσως ε, εγκληματίας, ε, παραβιάζεται το δίκαιο. Σε ό,τι αφορά τώρα τον Αμερικανό πρέσβη, ενδεχομένω, είπε και ο κύριος Φάρετς τα, τα σχετικά Ανέφερε γιατί τον πρέσβη, το οποίο ε, θεωρεί το Brexit είναι η αρχή μόνο, ότι το ευρώ πρέπει να καταρρεύσει και ότι όλα αυτά θα πρέπει να είναι στο μέλλον. Αλλά και εγώ θα ήθελα από πλευρά του ΕΛΚ να πω το εξή, ότι αν ε, έχουμε και θα πρέπει να καλωσορίσουμε εδώ πέρα έναν πρεσβευτή από την ΕΠΑ που αμφισβητεί το ευρώ και προβλέπει το τέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα μπορεί να διαπιστευτεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ απλά δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με έναν τέτοιον άνθρωπο και αγαπητοί συνάδελφοι, θέλει με πόλεμο να περάσει τα συμφέροντά του και ε, θέλει μία αδύναμη Ευρώπη. Και ο Ντόναλτ Τραμπ ε, θεωρούν ότι Κίνα και η Ευρώπη είναι οι μεγαλύτεροι οικονομικοί ανταγωνιστέ του και προσπαθεί να του αποδυναμώσει. Και θέλει λοιπόν μια ε, κατακριματισμένη Ευρώπη. Και γι' αυτό λοιπόν τι επόμενε εβδομάδε, μήνε και τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να δούμε κάποια βασικά πράγματα. Κατά πόσο είμαστε ενωμένοι. Αν μου επιτρέπετε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να πω και το εξή. Κοιτώντα την ιστορία των ΗΠΑ, την ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, μου έρχονται στο μυαλό ονόματα από το Ρούσβελτ και Τσέρτσιλ, πολιτικοί, οι, οποία, οι οποίοι πολέμησαν ε, πλευρό με πλευρό κατά της ε, αυταρχικότητας και των ε, πολλών εθνικών εγωισμών. Όχι τόσο πολύ α, να κοιτάμε τους εθνικούς, τα εθνικά συμφέροντα, αλλά να κοιτάμε τις αξίες. Ο Ρίγαν και, ο Ρίγκαν και η Θάτσερ ε, καταπολέμησαν τον κομμουνισμό. Όχι από εγωιστικούς λόγους για το ότι ήταν πιο σωστό για τη χώρα τους, αλλά γιατί ήταν το πιο σωστό για την κόσμο. Και τα δύο αυτά τζεύγια των πολιτικών πολέμησαν για την ελευθερία στον κόσμο. Και εγώ θα ήθελα και θα ευχόμουν να γινόταν το ίδιο σήμερα. Ο Ντόναλτ Τραμπ και η Τερίζα Μάη με, δυστυχώς ε, ε, προωθούν τον, τους εθνικά συμφέροντα, τον εθνικό εγωισμό, όχι τις αρχές για τον κόσμο. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο κόσμος μεταβάλλεται γρήγορα, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα στην Βαλέτα να αποσταλεί ένα σαφές μήνυμα, ένα χειρό μήνυμα, το οποίο το διευκρίνησε και ο Ντόναλτ Τάσκ στην επιστολή του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι προτεκτοράτο των είπα Αυτά τα λέει η Λεπέν και νομίζω ότι η Βαλέτα δεν μπορεί να είναι αυτό η Ευρώπη. Δεν είναι αυτό που χαρακτηρίζει τι αξίε μα και τι αρχέ. μα. Ευχαριστώ κύριε Βέμπερ για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες ο κύριος Πιτέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλοί πίστευαν ότι ο κύριος Τραμπ ήταν μια αστιότητα, ήταν ένα ανέκδοτο. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι πιστεύαμε. Εμείς δεν υποτιμούμε βέβαια την κατάσταση όταν το κάναμε αυτό στην ιστορία. Κάποιες προσωπικότητες έγιναν δικτάτορες και οδήγησαν σε πολέμους και σε αιματοχυσίες. Όπως είπε πολύ σωστά η κυρία Μογκερίνη η φιλία μας με τον Αμερικανικό λαό είναι αδιαμφισβήτητη. Είναι απαραίτητο και είναι μοναδική σταθερά αν θέλετε των αισθημάτων μας απέναντι στους υπόλοιπους λαούς και ο θαυμασμός μας επίσης για αυτό το οποίο έχουν υπάρξει στην ιστορία και για αυτό το οποίο είναι και σήμερα. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν είναι επώδυνο το να ακούει κανείς αυτές τις προτάσεις του Πρόεδρου Τραμπ που είναι μια επίθεση στον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό και στις αξίες μας. Μάνφρεντα ονοματίσουμε τα πράγματα σωστά. Αυτό που λέγεται travel ban απευθύνεται στους πολίτες ορισμένων χωρών δεν έχει καμία σχέση με τη διαχείριση των συνόρων και με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Είναι μια δημαγωγική ανοησία. Αυτή λέει είναι καλή, αυτή δεν είναι καλή. Με αυτού δηλαδή που έχει εμπορικές σχέσεις ο Τραμπ κανένα πρόβλημα. Με τους άλλους όμως υπάρχει πρόβλημα. Ας το πούμε όπως είναι λοιπόν τα πράγματα. Είναι μια επίθεση στην έννοια του ασύλου. Είναι μια επίθεση στην έννοια του κράτους δικαίου. Από ποιον, από τον άνθρωπο που θέλει να χτίσει τείχος στο Μεξικό, στα σύνορα με το Μεξικό. Νομίζω ότι αυτός ο ιός αποσταθεροποίησης και αναταραχής νομίζω είναι πολύ θλιβερό εγώ λέω στις αεροπορικές εταιρείες να μην υπακούσουν σε τέτοιου είδους μέτρα, να μην αρνηθούν στην επιβίβαση σε ανθρώπους οι οποίοι φύγονται από τις προτάσεις Τραμπ. Αυτό που είπατε για τον μελλοντικό σε εισαγωγικό <clears throat> πρέσβη ότι δεν θα είναι καλοδεχούμενος. Είναι λίγο περίεργο. Είναι ένας άνθρωπος που λέει ότι εγώ πάω εκεί για να βοηθήσω να καταστραφεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει στην κυρία Μέη μη βιάζεστε να λειτουργήσετε σαν δούριο ύπος για να καταστρέψετε από μέσα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, τα κράτη-μέλη το καθένα κάνει αυτό το οποίο επιθυμεί. Από την άλλη όμως καλό θα ήταν να υπάρξει ένα συντονισμό των πρέσβεων ε, στις Ηνωμένε Πολιτείες για το τι συμβαίνει εκεί και ακόμα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να συζητήσουμε το αν θα πρέπει να προσκληθεί ή όχι ο κύριος Τραμπ. Εγώ είμαι υπέρ της συνεργασίας με τους Αμερικανούς όπως και η Αντιπρόεδρος Μογκερίνη. Αν όμως ο Τραμπ δεν αλλάξει την γραμμή του τότε η πόρτα της Ευρώπης, η θύρα της Ευρώπης θα παραμείνει κλειστή για του συντηρητικού το λόγο έχει ο κύριος Σιάντ Κάμαλ. Ευχαριστώ. Έγινε μια μελέτη από το Ιστότο το Ίδρυμα Κάρτερ, που είναι ένα αξιοθέβαστο και το φιλελεύθερο ίδρυμα από το 1975 ε, κανένας Αμερικανός δεν σκοτώθηκε σε αμερικανικό έδαφος από υπήκο καμίας από αυτές τις 7 χώρες ε, που ε, είναι στα εκτελεστικά αυτά διδάγματα του Προέδρου Τραμπ. Όσοι λοιπόν πιστεύουν ότι θα πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη αλλά και ισότητα, να είναι όλοι ίσοι απέναντι προς τον νόμο, τότε πραγματικά ανησυχούν και δικαίως για αυτή την αυθαίρετη απαγόρευση που δεν πλήττει μόνο μουσουλμάνους αλλά και και χριστιανούς που φεύγουν να γλιτώσουν από τη δίωξη και το ε, θάνατο. Υπάρχουν επίσης κάποιες αντιφάσεις ε, το να είναι κανείς ένας καλός μουσουλμάνος, καλός πολίτης δημοκρατίας. Ε, αυτό ουσιαστικά είναι ένα χαρτί στα χέρια των ΤΑΕΣ και των εξτρεμιστών και τσιχαντιστών. Τα ίδια λένε και αυτοί όταν στρατολογούν απογοητευμένους, απελπισμένους νέους και νέες ως τρομοκράτες. Ό,τι και αν πιστεύουμε όμως εμείς, το γεγονός είναι ότι οι Αμερικάνοι ψήφισαν υπέρ ενός υποψήφιου που έλεγε αυτό που πίστευε. Και τώρα διαπιστώνω ότι έχουν ένα πρόεδρο που ε, κάνει πράξη τις υποσχέσεις του. Πρέπει λοιπόν αυτό να το δεχθούμε. Αυτός ο πρόεδρος έχει ως προτεραιότητες και ως πολιτικές αυτά ε, που είναι η συνέπεια της μεγάλης απογοήτευσης ε, που την διαπιστώνουμε όχι μόνο στη Βορειοαμερική αλλά και σε πολλές από δικέ δικές μας χώρες. Το κλινικό σώμα έχει χάσει την εμπιστοσύνη τους πολιτικούς και και κακήθεν του Ατλαντικού έχει χάσει την εμπιστοσύνη τους πολιτικούς ότι δεν μπορεί να ακούν, ε, δεν μπορούν ε, να αποδίδουν τα αποτελέσματα και τελικά οι πολίτες μας προσελκύονται από απλουστευτικές λύσεις ε, στα άκρα του πολιτικού φάσματος Εκφράζουμε τι ανησυχίε μα για τα εκτελεστικά διδάγματα του Πρόεδρου. Τραμπ. Ταυτόχρονα όμω, πρέπει να ε, ληφθούμε ότι όσο η ε, παγκοσμιοποίηση ε, είναι κάτι θετικό σε ό,τι αφορά τι επιχειρήσει και όχι σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους, αν δεν λαμβάνουμε υπόψη τη διαφορετικότητα, την κατανόηση και την αλλαγή και την ολοκλήρωση, τότε οι πολιτικέ θα συνεχίσουν να είναι παρόμοιε και οι πολιτικοί ε, στη Γαλλία, στην Ολλανδία και αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα κερδίζουν όταν εκφράζουν ακραίε απόψεις, λαϊκιστικές απόψει. το να λέμε ότι είναι ρατσιστικά ή ε, λαϊκιστικά όλα αυτά τα μέτρα, ε, αν δεν έχουμε να προσθέσουμε μία εναλλακτική εμείς, δεν θα είμαστε αξιόπιστοι. Πρέπει να διερωτηθούμε. Τι είναι πιο αποτελεσματικό η ένθερμη και θερμοκέφαλη αντίδραση ή η ψύχρεμη διπλωματία. Άλλωστε δεν ε, υπάρχουν ε, από το Κογκρέσο, ε, δεν έχει δοθεί έγκριση από το Κογκρέσο, δεν υποστηρίζεται αυτά τα διατάγματα και έτσι η Αμερική δεν θα γίνει ξανά μεγάλη, ούτε θα ενισχυθεί. Θα αποδυναμωθεί και η σχέση μας επίσης διατλαντική. Θέλω επίσης να σας πω ότι οι φίλοι πιο πολύ θα υποστηρίξουν ε, ε, κάποιους φίλους που μιλούν με τη λογική και την ψυχραιμία παρά τις κραυγές. Ε, Σας καλημερίζω όλους. Ο κύριος Φερχόφστατ έχει το λόγο από πλευράς της ομάδας των φιλελευθέρων. Has end his intervention and, uh, also... Ο κύριος Πιτέλα μίλησε και κάτι δεν καταλαβαίνω όμως από αυτά που είπατε κύριε Καμάλη. Καταρχάς είπατε ότι αυτό δεν γίνεται και μετά λέτε δύο φράσεις αργότερα αλλά πρέπει να το αποδεχτούμε γιατί είναι απο... εκλεγμένος. Όχι, δεν σημαίνει το ότι είναι εκλεγμένος ότι μπορεί να αντίκειται στις ανθρώπινες αξίες και τις αξίες των ΗΠΑ ακόμα και ένας εκλεγμένος πρόεδρος με την πλειοψηφία και δεν έχει πλειοψηφία τη λαϊκή ψήφου στη ΣΥΠΑ θα πρέπει να ακούει και να ακολουθεί το Αμερικανικό Σύνταγμα, το δικαστικό σώμα και εδώ ξεκινάω λοιπόν την παρέμβασή μου. Αυτό που λένε κάποιοι στη ΣΥΠΑ είναι ότι αυτό βοηθάει την ασφάλεια. Μα αυτό είναι νοησία ανοησία. Έχετε και τα δεδομένα μπροστά σα, τα αριθμητικά στοιχεία. Από το 1975 οι τρομοκράτε στη ΣΥΠΑ είναι από τρει χώρε. Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και Λίβανο. Καμία εξ αυτών δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των 7 χωρών. Και κανείς δεν ε, ήταν τρομοκράτης από τις χώρες αυτές. Πρόκειται για απλή και καθαρή διακριτική μεταχείριση. Διακριτική μεταχείριση σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο η θρησκευτική αυτή η απαγόρευση. Το θέμα είναι το, η τροφοδότηση του λαϊκισμού και του εθνικισμού. Αυτό κάνει η κυβέρνηση του Τραμπ. Και αυτό δεν είναι μόνο το γεγονό ότι διορίζει ω εκπρόσωπο του κ. Φαράτσο εδώ, αλλά διορίζοντα και τον Μάλακο ω πρεσβευτή και πιο σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε το Στίβ Πάνεν μέλος πλέον του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας τον είπα. Έναν άνθρωπο ο οποίος ανοιχτά βγαίνει και διακηρύττει ότι θέλουν τα αδεξιά κινήματα να ξεφορτωθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και, και εδώ είναι και κάθονται η πέμπτη στήλη. Γιατί ο κύριος Φάρατς συνεργάζεται μαζί του. Τον βλέπει σε τακτική βάση. Για ένα και μόνο σκοπό για την καταστροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα έτη. χωρίς να σκέφτεται αγαπητοί συνάδελφοι ένα πράγμα. Ότι είναι μεγάλο το ρίσκο το να γνωστηριστεί κανεί στον εθνικισμό και τον λαϊκισμό στην Ευρώπη. Το ζήσαμε αυτό τα ζήσαμε αυτά στον 20ο αιώνα και είδαμε. Και ήταν άνθρωποι που πίστεψαν ότι ο αιωνα και ειδαμε και ηταν ανθρωποι που πιστεψαν οτι ο λαικισμος και ο εθνικισμό ήταν η λύση για την ήπειρό μα. Και ζήσαμε τι πιο φρικτέ φρικαλαιότητες. 20 εκατομμύρια ζωέ κόστησε ο εθνικισμό στην Ευρώπη. Και δεν υπάρχει ούτε μία οικογένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχασε κάποιον από την οικογένειά του, κάποιον πατέρα, αδερφό, παππού κόρη θύμα αυτού του εθνικισμού και του λαϊκισμού και γι' αυτό λοιπόν δημιουργήσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξεπεράσουμε τα πράγματα αυτά, για να υπάρξει μια ήπειρος ειρήνης και πιστεύω αυτό που βλέπω στην παρούσα φάση είναι κάτι που δεν κάνει κανονικά ένα Αμερικανό πρόεδρο, ο Ρούσβελτ, που ήταν να είναι ο ηγέτη του ελεύθερου κόσμου. Δεν βλέπω έναν Αμερικανό πρόεδρο που θέλει να είναι Τέτοιο πρόεδρο, Τώρα βλέπω έναν πρόεδρο ο οποίος θέλει να είναι ο ηγέτη τη καταπολέμησης τη ελευθερία του ελεύθερου κόσμου και είναι πραγματικά υπεραξιακή στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αγαπητέ κύριε πρόεδρε μου. Η απόφαση μόνο έχουμε να πάρουμε τον Πούτιν ή την Ευρώπη, τον Τραμπ ε, μια εθνικιστική, λαϊκιστική άποψη που θέλει να μας καταστρέψει. Έχουμε την απειλή του εξτρεμισμού και έχουμε και εδώ και ένα μάτσο άτομα που θέλουν να μας καταστρέψουν εκ των έσω. Ένα πράγμα λοιπόν μπορούμε να κάνουμε, να ενωθούμε και να αντισταθούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ελπίζω ότι στη Βαλέτα όχι μόνο την επιστολή θα έχουμε που την υποστηρίζω την επιστολή του Πρόεδρου Τάσκ. Ελπίζω να μην έχουμε μόνο αυτό. Ελπίζω μια φορά όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες να μπορέσουν να ενώθησουν την γροθιά τους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να πολεμήσουν αυτό το μάτσο τους ε, λαϊκιστές που θέλουν να μας καταστρέψουν. Ευχαριστώ κυρία Τσίμερ για την ΚΟΥΕΝΤΖΙΕΛ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα δεν είναι η πρώτη ούτε τελευταία φορά σήμερα που θα συζητήσουμε την πολιτική των Πολιτειών και ιδίω τη κυβέρνηση ε, Τραμπ. Θα μα απασχολήσει και στο μέλλον η πολιτική Τραμπ. Κυρία Μογκερίνη, είπατε ότι υπάρχει μια ε, σχέση χρονική με την ε, με τα διατάγματα ε, του Τραμπ. Ε, είπατε 27 Ιανουαρίου έγινε αυτή, βγήκε αυτό το διάταγμα κατά της ε, εισόδου μουσουλμάνων στις ΗΠΑ. Είναι, όμως υπάρχει ένα σύστημα, υπάρχει ένας λόγος που γίνονται όλα αυτά. Γιατί Έχουμε συζητήσει και για τις ζωές που χάθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης ε, στη ναζιστική Γερμανική αλλού. Ε, όταν έγιναν κάποιες τέτοιες δηλώσεις ε, προς τον Τράπο, ο Τραμπ είπε στο συγκεκριμένο ότι δεν είναι καλός ηθοποιός. Εμείς πρέπει τώρα να αποδείξουμε ότι το δικό μας σύστημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει να προσφέρει κάτι αναλλακτικό, κάτι διαφορετικό από αυτήν ε, την ε, έλλειψη σεβασμού προς τον άνθρωπο. Πρέπει να αποδείξουμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι και εσείς ε, μιλήσατε και είπατε σε ένα tweet ότι είμαστε ασφαλείς για τους μετανάστες σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως δεν ισχύει ούτε αυτό. Αυτό μπορούμε εμείς ε, να το αποδείξουμε. Εμείς πρέπει πάντως να σταθούμε απέναντι στον τραπ. πρέπει να ευθύσουμε μια αλληλέγγυα μεταναστευτική πολιτική ε, και οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται εδώ να βρουν ένα καταφύγιο όταν φεύγουν από την ε, τρομοκρατία και από την εγκληματικότητα. Και αυτοί που έρχονται εδώ δεν είναι ούτε εγκληματίε ούτε τρομοκράτε. Θέλουν να, να δράσουν μαζί μα από κοινού κατάλληλων αυτών τι θα γινόταν μετά το 1945. Εδώ γεννήθηκε ξανά η δημοκρατία. Ξέρουμε ότι ε, η ναζιστική δημοκρατία, η ναζιστική Γερμανία σκόρπισε όλεθρο μέχρι τότε. Αν όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι ε, δεν είχαν έλθει εδώ μετά, πού θα βρισκόμασταν και θα πρέπει να μην παίξουμε τα παιχνίδια αυτά που ακούγονται. Θα πρέπει να αντεπιτεθούμε και μάλιστα με αυτό που μπορούμε καλύτερα να κάνουμε και να αποδείξουμε ότι δηλαδή έχουμε να προσφέρουμε κάτι καλύτερο και μαζί με τους Αμερικανούς πολίτες θα πρέπει να συνεργαστούμε με αυτούς που έχουν κοινέ αξίες με εμάς. Αυτό που μου έδωσε ελπίδα σήμερα είναι ότι αμέσως μόλις ανέλαβε καθήκοντα και τις επόμενες ημέρες ο Τραμπ παντού στον κόσμο και ιδίως στη ΣΥΠΑ χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες στράφηκαν κατά αυτής της εικόνας και αυτού του στερεότυπου, όχι μόνο κατά της δεκτικής μεταχείρισης σε βάρος των γυναικών, γιατί το θέμα είναι αξιοπρέπεια, ανθρώπινη, ο σεβασμός προς τον άνθρωπο, ε, κανένας αποκλεισμός, καμία δεκτική μεταχείριση, ανεξαρτήτως φύλου, ε, κτλ. Αυτό ακριβώς πρέπει και εμείς να επιβάλλουμε. Πρέπει να καταπολεμήσουμε την ιδεολογία Τραμπ και των ίδιων θα πρέπει εμείς να βοηθήσουμε για περισσότερη ασφάλεια. Παραδείγματο χάρη κλείνοντα όλου του πυρηνικού σταθμού που υπάρχουν και κάποιοι στη Γερμανία. Αυτά πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ κυρία Κέλλερ για την ομάδα των Πρασίνων. Thank you. Ευχαριστώ. Ο 45ος λοιπόν πρόεδρος ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και της δημοκρατίας. Αυτή η απαγόρευση για επτά χώρες δεν είναι κάτι το οποίο προωθεί την ασφάλεια ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα απλό ε, μέτρο διάκρισης εις βάρος των μουσουλμάνων. Δεν φύγει βέβαια όλους τους μουσουλμάνους, παρόλα αυτά στοχεύει εναντίον των μουσουλμάνων λόγω της θρησκείας τους. Ποιος θα πίστευε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί. Ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι η ελευθερία και τα δικαιώματα τα οποία θεωρούνται δεδομένα σε διεθνές επίπεδο θα εξανεμιζόντουσαν τόσο γρήγορα. Αυτό δείχνει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποθάνει η φιλελεύθερη δημοκρατία μέσω ενός προεδρικού διατάγματος. Νομίζω ότι δυστυχώς το αμερικανικό όνειρο δεν έχει αφήσει τίποτα, εξαφανίστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Βλέπουμε ότι τα δικαιώματα, οι ελευθερίες που θεωρούμε δεδομένα, μόνο δεδομένα δεν είναι. Πάντα πρέπει να δίνει μάχη κανείς για αυτά σε καθημερινή βάση και σε κάθε στιγμή. Ε, η δημοκρατία φυσικά είναι εγγεγραμμένη στη συνταγματική μας τάξη, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Πρέπει να δίνουμε μάχη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να δουλεύει κανείς για αυτά καθημερινά. Στην Ευρώπη είμαστε υπερήφανοι ότι ζούμε σε μια ένωση δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Δεν αρκεί όμως το να το αναγνωρίζουμε αυτό. Και εμείς δυστυχώς βάζουμε περιορισμού στα σύνορά μας. Και εμείς σηκώνουμε φράγματα. Και εμείς εδώ μερικές φορές αναφερόμαστε σε διακρίσεις λόγω προέλευσης, λόγω θρησκείας κλπ. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς για τους εαυτούς μας. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι και κυρίως οι κυβερνήσεις των κρατών μελών θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν με ποιους είμαστε. Είμαστε με το μίσος, είμαστε με την καταδίκη ή είμαστε με τη δημοκρατία και με τις γέφυρες. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να συνέλθουμε, να λύσουμε την οικονομική κρίση η οποία οδηγεί στην ανεργία των νέων Πρέπει να συντονίσουμε τις εξωτερικές μας πολιτικές και να γίνουμε πρωταθλητές του διεθνούς δικαίου. Γιατί δεν υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι που θα το έκαναν αυτό. Πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο μας και στον Ηνωμένο Εθνό και στην προστασία του κλίματος. Ας καταστήσουμε λοιπόν την Ευρώπη το αντίθετο του Τραμπ στην ελευθερία, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο κράτος δικαίου, στην γενεοδορία. Ας δείξουμε την δικαιοσύνη μας. Ας δείξουμε το πάθος μας για τη δικαιοσύνη. Να μην μιλάμε όμως μόνο για αυτά, να το αποδεικνύουμε σε καθημερινή βάση το αγαλμά της ελευθερίας το χάρισε η Γαλλία στη νέα της αδελφή της Ηνωμένε Πολιτείες. Νομίζω ότι το σύμβολο αυτό της ελευθερίας θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε άλλα μέρη όπως τη Λαμπεδούσα, όπως τη Μιτιλίνη όπου όλοι ξαφνικά φτάνουν εκεί γεμάτοι ελπίδα. Πρέπει λοιπόν να πολεμήσουμε για τα δικαιώματά τους, για τα δικαιώματα των γειτόνων μας, για τα δικαιώματα αυτών οι οποίοι παλεύουν για όλους ανεξαρτήτως της καταγωγής τους, της θρησκείας, της προέλευσης, ε, του γενετήσου προσανατολισμού. Η Ευρώπη χτίζει γέφυρες, δεν χτίζει τείχη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φαράζ. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι όλοι είστε πάλι αναστατωμένοι εδώ πέρα σήμερα το απόγευμα. Δεν αμφιβάλλω ότι τα γεγονότα στη ΣΥΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες ήταν ε, ένα βαθύ σοκ για σας και ίσως έχετε δίκιο γιατί βλέπετε τι έχει συμβεί εδώ. Κάποιος ε, ο οποίος ε, μπήκε σε εκλογές, πήρε το αξίωμα και μέσα σε μία εβδομάδα είπε ότι θα τηρούσε το Εκλογικέ τους υποσχέσεις. Πραγματική και ειλικρινή ε, αυθεντική δημοκρατία, αντίθετα με το σύστημα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου μη εκλεγμένοι, όπω η κυρία Μογκερίνη εδώ, έχουν το δικαίωμα να προτείνουν νομοθεσία. Φαντάζομαι σε σοκάρει πάρα πολύ να δείτε τι κάνει μια αυθεντική δημοκρατία, ένα αυθεντικά εκλεγμένο ε, από δημοκρατικό σύστημα. Φαντάζομαι ότι είναι σοκ. Συγγνώμη, σχόλια εκτός μικροφώνου. Κοιτάξτε, πρέπει να σεβαστείτε το Κοινοβούλιο, πρέπει να σεβαστείτε επίσης τις θεσμικές αρμοδιότητες των ε, επιτρόπων. Όχι μόνο γιατί πρέπει να δείχνει κανείς σεβασμό, αλλά για να αναγνωρίσουμε και την καλή πρόθεση της Αντιπροέδρου και υπά της εκπροσώπου της, κυρίας Μογερίνη. Μάλιστα και από θεσμικό σεβασμό προς την αλήθεια κύριε Πρόεδρε θα καταλαβαίνετε και θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η μία εκλεγμένη κομισιόν είναι η μοναδική που έχει το δικαίωμα να προτείνει νομοθεσία και αν έχω λάθο και αν το κάνω λάθο, να μετρώ έξω από το κοινοβούλιο αυτό εδώ και τώρα σήμερα το απόγευμα. Κύριε Φαράζ, Κοιτάξτε, παρακαλώ σα ζητώ να δείξετε για μια ακόμη φορά σεβασμό, τίποτα άλλο. Συνεχίστε παρακαλώ. Oh, Θα επιδείξω σεβασμό, να είστε σίγουρο, αλλά και εσεί να επιδείξετε σεβασμό για το δικαίωμα του ηγέτη ενό πολιτικού κόμματο, μια πολιτική ομάδα που έχει κερδίσει τι εκλογέ του 2014, τι ευρωεκλογέ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και μου φαίνεται ότι με όλη την τροτική κατά του Κραμπ που προέρχεται από παντού, αυτό που ακούμε είναι το εξή. Η πραγματική φύση του ευρωπαϊκού έργου που είναι πραγματικά αυθεντικό αντιαμερικανισμό. Ο Τραμπ έχει ως κίνητρο την προστασία των ΗΠΑ από, τον Ισλαμικό, από την Ισλαμική τρομοκρατία. Ενώ αυτό που συνέβη εδώ στην αίθουσα αυτή και στις κυβερνήσεις της Ευρώπης είναι ότι τους καλωσορίσατε τους ανθρώπους αυτούς στα σπίτια σας, μέσα στη φωλιά σας για μια στιγμή μόνο να κοιτάξουμε το εξή γεγονό μέσα από τι υπερβολέ και μέσα από την ιστερία ότι το μοναδικό που έκανε ο Ντόναλτ Τραμπ είναι ότι πήρε 7 χώρε που έχουν εντοπιστεί από τον πρόεδρο Ομπάμα ως επικίνδυνες για τις ΗΠΑ. Ο Ομπάμα ήδη είχε περάσει μια διαδικασία ελέγχου. Και αυτό που έκανε ο Τραμπ είναι για 90 μέρε είπε α εξετάσουμε αυτόν τον έλεγχο, να δούμε κατά πόσον αρκεί. Να σα ρωτήσω εσά κύριε Φερχόφστατ και όλου του υπόλοιπου με, τις ψευδείς, με την ψευδή αγανάκτησή σα. Πού ήσασταν το 2011 που ο Ομπάμα απαγόρευσε από κάθε κοινό να μπει στη ΣΥΠΑ για ένα χρόνο. Γιατί δεν ακούω καμία κριτική για τη Σαουδική Αραβία, για τον Μπαχρέιν, το Κουβέιτ που αρνήθηκαν να δεχτούν έναν, έναν μόνο πρόσφυγα ή εκτοπισμένο από τη Συρία. Και πώς είναι δυνατόν την ημέρα του ολοκαυτώματος, την προηγούμενη Παρασκευή, ούτε ένας από εσά δεν επέκρινε όσους ε, δεν επιτρέπουν στους Ελληνούς Εβραίους να πάνε στη χώρα τους να πάνε στη χώρα τους για διακοπές. Πού, τι υποκρισία είναι αυτή. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε ενδεχομένω είναι να είμαστε κάπως πιο επικοδομητικοί. Όλοι μας εδώ λέμε και διτεινόμαστε ότι είμαστε δημοκράτες. Να η ευκαιρία να το αποδείξουμε. Ας καλέσουμε τον πρόεδρο Τραμπ να έλθει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι βέβαιος ότι ως δημοκράτες θα συμφωνήσετε όλοι. Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι ανοιχτό ο διάλογο με τον εκλεκτέντα πιο ισχυρό άνθρωπο του κόσμου. Και αν το απορρίψετε αυτό ως πρόταση θα αποδείξετε ότι είσαστε οι αντιδημοκράτες που πάντα πίστευα ότι είσαστε. Καλώς σας ευχαριστώ κύριε Φερχώσταρτ. ΔΕΧΡΕΦ ΙΕΝΕΦ. President, Mr. Κύριε Πρόεδρε, πρόσφατα ο κύριος Τούσκ είπε ότι είπα είναι απειλή για την Ευρώπη όσο το Ισλαμικό κράτος μήπως, μήπως πάσχει από κρίση πανικού κύριος Τούσκ και έχει χάσει την αίσθηση της πραγματικότητας. Προσωρινά απαγορεύσει την είσοδο κύριος Τραμπ σε επικούς χωρών που και ο προκάτοχος του κύριος Ομπάμα, το είπε και ο κύριος Φάρατς ήδη, τις είχε ε, χαρακτηρίσει χώρες ε, που δημιουργούν κίνδυνο για την Αμερικανική δημόσια ασφάλεια. Είναι απόλυτα έγκυρο το να ε, καθεωρι... καθιερώνονται συνοριακοί έλεγχοι. Εδώ εμείς βλέπουμε τα αποτελέσματα ε, των αποτυχημένων ε, συνοριακών ελέγχων και είδαμε τις επιθέσεις ε, στη, στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες, στη Νίκαια, στο Βερολίνο. Είδαμε πόσες ζωές χάθηκαν και πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο Τραμπ λέει ότι είναι χάος η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει δίκιο γιατί περί αυτού ακριβώς πρόκειται. Η καταγραφή κατά του Προέδρου Τραμπ δεν είναι τίποτα άλλο παρά καθαρή υποκρισία. Το και ο Φαράτς. Πού ήταν ε, οι διαμαρτυρίες όταν οι Ισραηλινοί αποκλείονταν από τις ίδιες Ισλαμικές χώρες που τώρα τις αποκλείουν, είπα, πρέπει να ντρέπεστε που θέτεται σε κίνδυνο τις ζωές ανθρώπων, πολιτών της Ένωσης, ε, λόγω των ανελειπών συνοριακών έλεγχων. Καλό την Κομισιόν, καλό τον κύριο Τούσκ να ακολουθήσει το παράδειγμα του κύριου και να εγκαθιδρύσει εθνικού συνορικέ ελέγχου για να κρατήσει έξω του τζιχαντιστέ και όχι μόνο από τι 7 χώρε που έχει αναφέρει ο ο Τραμπ, αλλά και από πολλέ άλλε χώρε που είναι υπεύθυνε για αυτά τα παράνομα κύματα λαθρομεταναστών. Ευχαριστώ. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Νάιτζελ Φαρέτς, ένα μέλος των σε κάθισε πίσω του με ένα α, μήνυμα όλη την ώρα, με ένα, με ένα φλάδιο. Ελπίζω να γίνει κάτι, να επιταρχηθεί αυτό το μέλος ή τα να πάω και εγώ να κάτσω κάπου αλλού. Και εγώ να κάνω το ίδιο. Κύριε Έθεριτζ, κύριε Έθεριτζ, στείλαμε τους κλητήρους να πούν στον συνάδελφό σας ότι δεν έπρεπε να σηκώσει την ταμπέλα που σήκωσε. Για τους μη εγγεγραμμένους ο κύριος Παπαδάκης. ενάμιση λεπτό παρακαλώ. Η επιλογή Τραμπ εκφράζει ανακατατάξει ανάμεσα σε μερίδες του κεφαλαίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι απαράδεκτες απαγορεύσεις και τα μέτρα καταστολής της διακυβέρνησης Τραμπ συνιστούν επικίνδυνη εξέλιξη βάζουν στο στόχαστρο εκατομμύρια μετανάστες και πρόσφυγες μεγάλα θύματα του καπιταλιστικού συστήματος που διαχειρίζεται και η διακυβέρνηση τραμπ. στόχος η μέγιστη κερδοφορία των αμερικάνικων επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος των αμερικανών εργαζομένων. οι κινήσεις οικονομικού προστατευτισμού των ΗΠΑ που συγκεντρώνουν δυνάμεις στην αντιπαράθεσή τους με την κίνα επιχειρώντας προσέγγιση με τη ρωσία οξύνουν τις αντιθέσεις δρομολογούν ανακατατάξεις. το brexit η στήριξη των λεγόμενων ευρωσκεπτικιστών αποτελούν απάντηση μερίδας του κεφαλαίου στην ευρώπη που δεν κερδίζει όσα υπολόγιζε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ένωσης αξιοποιώντας κιόλας και τη λαϊκή δυσαρέσκεια. η συνοχή της ευρωπαϊκής ένωσης και της ευρωζώνης θα δοκιμαστούν. πιθανός είναι και ο σχηματισμός άλλων συμμαχιών εξίσου αντιδραστικών με την ευρωπαϊκή ένωση οι λαοί να απορρίψουν κάθε συμμαχία του κεφαλαίου να βαδίσουν τον δρόμο των δικών τους συμφερόντων για άλλη νέα οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας αποδεσμευμένη από τις αλυσίδες των λικοσυμμαχιών τύπου ευρωπαϊκής ένωσης και νάτο. E eh, Je Για την απάντηση, κυρία σα ευχαριστώ και θα μιλήσω αγγλικά νομίζω γιατί να είναι καλύτερα αυτό. Νομίζω ότι ο σεβασμό του ρόλου τη ε, απόστολη και ιδιαίτερω ε, στην περίπτωσή μου ε, τη θέση, τη είπα εκπροσώπου τη Κομισιόν είναι και σημάδι και ένδειξη σεβασμού προ το Κοινοβούλιο γιατί με, γιατί με ανέθεσαν στη θέση αυτή το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών που είναι εκλεγμένοι, αλλά βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη σύγχυση και στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε κάποια τμήματα του Ηνωμένου Βασίλειου. Η ΕΠΑ είναι μια μεγάλη χώρα, μια μεγάλη δημοκρατία. Η, η Αμερική θα πρέπει να αντιμετωπίσει τους διχασμούς της και να κάνει τις συζητήσεις που έχει να κάνει. Και ξέρω ότι ως Ευρωπαίοι είμαστε ειδικευμένοι να οικειοποιούμαστε κάθε κρίση. Νομίζω ότι είναι σαφές όμως ότι αυτή η κρίση είναι κρίση της Αμερικής και θα πρέπει οι Αμερικανοί να την επιλύσουν με όποιο τρόπο μπορούν. Ξεκινώντας από τις επικίνδυνες πολλώσεις και ατυχασμούς που βλέπουμε στο αμερικανικό πολιτικό και οικονομικό σκηνικό. Αλλά είμαι αισιόδοξη. Πιστεύω ότι οι Αμερικανοί φίλοι, μου, φίλοι μας θα βρουν τον τρόπο να ξεπεράσουν τις κρίσεις αυτές και τις τριβές αυτές και θα εξακολουθήσουν να αποτελούν τη μεγάλη χώρα που είναι και που θα συνεχίσουν να είναι. Εμείς τι έχουμε να κάνουμε. Εμείς δεν ε, θα λύσουμε τις ε, τρέχουσες αμερικανικές ε, πολλώσεις και τους διχασμούς, αλλά θα πρέπει να βεβαιώσουμε εκ νέου τις δικές μας αξίες, τις δικές μας πολιτικές και να είμαστε πιστοί σε αυτές. Και έχετε απόλυτα δίκιο όσοι το τονίσατε αυτό. Θα πρέπει να είμαστε πραγματικά α, πιστοί στις αρχές μας και στις αξίες μας. Να είμαστε λοιπόν δυνατοί και να επιδείξουμε ηγεσία. Και αυτό γιατί μπορεί να έχουμε χάσει σε κάποια θέματα ένα σημαντικό εταίρο, αλλά αυτό καθιστά την ηγεσία από πλευρά μα ακόμα πιο σημαντική και επίκαιρη και πραγματικά απαραίτητη. Σε όλο τον κόσμο λοιπόν στην περιοχή μας ε, και πολύ μακριά από εδώ ο κόσμος αντενίζει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, τώρα, ο σημείο αναφοράς σε ό,τι αφορά την πολυμέρεια, σε ό,τι αφορά το ελεύθερο και το δίκαιο εμπόριο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το σεβασμό, που για μας αποτελεί τη βάση όχι μόνο των δοσμικών σχέσεων, αλλά και των ανθρωπίνων σχέσεων, σε ό,τι αφορά τον ουμανισμό την ανθρωπιά μας, αν θέλετε. Αλλά έτσι είμαστε εμείς οι Ευρωπαίοι. Κάποιες φορές δεν είμαστε αρκετά περήφανοι για το ποιοι είμαστε και για το τι μπορούμε να γίνουμε. Και θα ήθελα να κλείσω λέγοντας το εξής. Κάποιοι μεγάλοι Αμερικανοί φίλοι μας πριν από κάποιους μήνες εδώ πέρα μας επενθύμησαν στις Βρυξέλλες ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να πιστεύουν στον εαυτό τους όσο πιστεύουν και όλοι οι φίλοι τους στον κόσμο σε εμάς και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα και η στιγμή να εκπληρώσουμε το δυναμικό μας και να μπορέσουμε να αποτελέσουμε το ισχυρό σημείο αναφοράς που χρειάζεται όλος ο κόσμος και όλη η περιοχή μας, όλος ιδιαίτερος. Και σκεφτόμουν το παράδοξο. Θα έχουμε ένα πρωθυπουργό της ε, Λιβύης εδώ αύριο. Αυτή η πρόσκληση προήλθε, μάλλον έγινε πριν ε, ληφθεί η εκτελεστική απόφαση απαγόρευσης εισόδου. Όταν ε, κανείς ε, ορθώνει τύχη, μπορεί να έχει την αίσθηση ότι είναι πιο ασφαλής, αλλά ουσιαστικά αποστερεί τον εαυτό του από οποιαδήποτε ευκαιρία. Εμείς οι Ευρωπαίοι δεν είμαστε έτσι και θα συνεχίσουμε να είμαστε πιστοί στις αξίες μας και στη λειτουργία μας, η οποία είναι συνεργασία και όχι αντιπαράθεση. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό και να το ακολουθήσουμε όσο εδώ και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Αντιπρόεδρο Μογκερίνη, ευχαριστώ και όσους όλους πήραν μέρος στη συζήτηση. Έχει